Ε, προασπιζόμαστε την ελευθερία και την ε, δίκαιη εκδίκαση υποθέσεων σε όλες τις χώρες και στην Τουρκία. Ήθελα να σας πληροφορήσω ότι στην μεικτή με, την Τινησία μια αντιπροσωπεία με τον κύριο Μοχάμπετ Φαντές Μπεν Ομράν κάνει μια επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω τον κύριο Μπεν Ομράν και τα μέλη της αντιπροσωπείας του και θα ήθελα να τονίσω την σημασία που αποδίδουμε σε αυτή την επίσκεψη. Να προχωρήσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Πρώτα απ' όλα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων